Ιουνίου από τις 9 έως τις 1 και μισή και από τις 3 έως τις 19.00 ε, και από τις 21.00 έως τις 24.00. Η μερίσια διάταξη έχει τυπωθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, την προσοχή σας. Λίγη συνεδρίασή μας. Γεια σας.